Μισό λεπτό ε, διακόπτει ο πρόεδρος, κυρία Φερέιρα. Muito obrigado, Sr. Presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συζήτηση με τον ε, Πορτογάλο Πρωθυπουργό στις αρχικές ε, παρεμβάσεις των Προέδρων των διαφόρων ομάδων αυτές οι παρεμβάσεις ξεπέρασαν κατά πολύ το χρόνο που είχε οριστεί. Η πρώτη παρέμβαση της δικής μας ομάδας στήρισε το χρόνο. Εάν πρέπει να, να... να αφαιρέσετε ε, χρόνο από κάποιου ανθρώπου, αυτή η διαδικασία που είχε συμφωνηθεί αλλά δηλαδή δεν τηρήθηκε, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρέσετε το χρόνο από το SDA από τις ομάδες που ξεπέρασαν τις παρεμβάσεις, το χρόνο παρέμβασής τους. Εμείς στηρίσαμε το χρώμα μας, μας στηρίσατε χρόνο στη συζήτηση στο Catch αλλά αυτό δεν σύμφωνε με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί και δεν θέλουμε να αφήσουμε, να, δεν θέλουμε να μην διαμαρτυρηθούμε, θέλουμε δηλαδή να διαμαρτυρηθούμε για αυτή τη διαδικασία που δεν είναι δίκαιη. Κύριε Φεραίρα, δώσαμε το λόγο αναλογικά σε όλες τις ομάδες. Ε, νομίζω ότι έγιναν σεβαστές όλες οι παρεμβάσεις. Τι να σας κάνω. Εσείς μπορεί να λέτε όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Μπορείτε να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε, αλλά οι υπολογισμοί έγιναν από τις υπηρεσίες με μαθηματικό τύπο. Ε, δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται μόνο από το ποια είναι η κατάσταση στην Αθήνα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Δημοκρατίας ε, μου διαβίβασαν το αίτημα άρσης ε, της ασυλίας του κ. Γεωργίου Κίρτσου για να ξεκινήσει η διαδικασία στο πρωτοδικείο της Αθήνας. Με βάση τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, το αίτημα αυτό διαβίβασε στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου την καθήλυν αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα την ψηφοφορία. Ε, ξεκινάμε με την ψηφοφορία για τις κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε.